Άρχεται η συνεδρίαση. Μετά από την διακοπή τη συνεδρίαση χθε το βράδυ, επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διαταξή μα είναι η παρουσίαση από το Συμβούλιο του Σχεδίου του Γενικού Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2010. Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω